Ακολουθεί η ψηφοφορία <clears throat> για το ψήφισμα τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών σε ό,τι αφορά την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών. Καταρχήν, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 6 κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 10 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Τροπολογία 3. Θέτω σε ψηφοφορία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 16 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι Κατά. Απόχες. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτό. Παράγραφος 18 ψήφι Κατά. Απόχες θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την παράγραφο 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Παράγραφο 24. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 27 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε με χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του εισαιτιολογικής σκέψης ε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται πράγματι. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Λατινική. Λατινικό Β. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. Το ψήφισμα ως σύνολο και όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ακολουθεί η ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα σε σχέση με την πολιτική επίλυση του προβλήματος της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας. Κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων που αντικαθιστά όλα τα άλλα ψηφίσματα. Τροπολογία 9 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική κλίση. Έναξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 11. Ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12. Έναρξη ψηφοφορία. Για την τροπολογία 12. Αν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία τώρα. Απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την παράγραφο 4 σε δύο τμήματα και τα δύο με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Αν ψηφίσατε όλοι, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 6. Πέρας. Απορρίπτεται. Η παράγραφο 8. Να ψηφίσουμε υπέρ. Για την παράγραφο 8. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη. Αν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 11. Αλλά με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία περιθμών 7. Και πάλι με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ παρακαλώ. Για την τροπολογία 13. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος που έχουν υποβάλει έξι πολιτικές ομάδες για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Να ελέγξουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην παράγραφο 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε τμήματα. Τρία τμήματα. Όλα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα για την παράγραφο 9 λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορίας. για την ξεχωριστή ψηφοφορία για το άρθρο 7. Την παραλείψατε. Ναι, όχι, μόλις ψηφίσαμε, λέει η Πρόεδρος. Εγκρίθηκε. We have a vote open. Ψηφοφορία, λοιπόν, για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 9. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην παράγραφο 9, δεύτερο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο τρίτο τμήμα. Α, συγγνώμη, καταπίπτεται το τρίτο τμήμα. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμό 3. Υπέρ. Κατά. Για την τροπολογία 3 δεν υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία, δεν προβλέπεται. Για την τροπολογία λοιπόν υπαριθμό 3 υπέρ. Κατά. So that we are clear. Για να διευκρινίσω την κατάσταση, συνάδελφοι, το, το τρίτο τμήμα της προηγούμενης παραγράφου κατέπεσε. Δεν το ψηφίσαμε λοιπόν τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία υπεριθμών 3 για την παράγραφο 10 του κυρίου Χάνς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. κυρία Κόλ, Βόρτμαν Κόλ. Πρόεδρε, το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Όχι, απορρίφθηκε, λέει η Πρόεδρο. Συμφωνείτε, γι' αυτό λοιπόν κατέπεσε το τρίτο τμήμα και γι' αυτό περάσαμε στην επόμενη ψηφοφορία. Να προχωρήσουμε με την παράγραφο 13. Τροπολογία 4, με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας, λοιπόν. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην παράγραφο 18. Με ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ για την παράγραφο 18. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το επόμενο θέμα είναι ψηφοφορία για τις προτάσεις ψηφίσματος για την κύρωση και εφαρμογή των ανθεωρημένων συμβάσεων της ΔΟΕ. Θα ψηφίσουμε ένα, μια κοινή πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων ομάδων. Δεν έχουμε τροπολογίες. Να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος για, μάλλον η ψηφοφορία για έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος για παγκόσμια διάσκεψη του ΦΑΟ για την επιστημική ασφάλεια πέντε πολιτικών ομάδων και θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας για το κοινό αυτοψήφισμα. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι.